Okay, colleagues, I suggest that we start with our meeting. Could you please take your... Παρακαλώ καθίστε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. I open the meeting. The first time, uh, first item of our agenda. Λοιπόν, πρώτο σημείο. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης, σχεδίου ημερήσιας διάταξης. Thank you. Uh, the draft agenda was emailed. Σας απεστάλλει με email στις 2 Απριλίου η ημερήσια διάταξη, είναι στους φακέλους σας. Προσέξτε, έχουμε κάνει μια μικρή αλλαγή. Σημείο 7, η γνωμοδότηση του κ. Σταυρακάκη. Θα ακολουθήσει το σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης. Και το σημείο 5, γνωμοδότηση Κάταλιν, θα πάει μετά το 6. Σημείο 2 Ανακοινώσεις Προέδρου. Έχουμε διερμηνία, έχουμε όλες τις καμπίνες εκτός από Δανέζικα. Ε, βγαίνει και στο διαδίκτυο, εκπέμπεται στο διαδίκτυο με web stripping. Η συνεδρίασή μας, τρία είναι έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων μας. Έχει τα πρακτικά της συνεδριάσεως της 20 ε, Μαρτίου του 2012. Σας απεστάλησαν στις 17 Απριλίου με email τα πρακτικά, δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ας θεωρηθούν ως συγκεκριμένα τα πρακτικά αυτά. Σημείο 4. Η ειδική έκθεση υπαριθμών 16 του 2011 οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για Σλοβακία, Λιθουανία και Βουλγαρία για αφοπλισμό ε, διαφόρων πυρηνικών αντιδραστήρων Μαρινέσκου ε, η στον κύριο Φαζάκα θα δώσω του ελεγκτικού συνεδρίου τον εκπρόσωπο το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμα μέλη. Καταρχάς εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού που έβαλε στο σημείο αυτό τη ημερήσια διατάξεω την ειδική έκθεση του Ελεκτικού Συνέδριου για την οικονομική βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για τον αφοπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων ει Βουλγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερος τον κύριο Μαρινέσκου και να εκφράσω την εκτίμησή μου σε αυτόν και στην ομάδα του διότι εφοσιώθηκαν σε αυτό το πολύ σημαντικό θέμα και ήταν πάρα πολύ πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μας. Θα γνωρίζετε ότι η πυρηνική ασφάλεια και ο φοπλισμός, η επεγκατάσταση αυτών των μονάδων ε, είναι κάτι που γίνεται όλο και πιο σημαντικό σε θέμα διότι ένα τρίτο από τους 143 πυρηνικούς αντιδραστήρες που λειτουργούν τώρα στην Ευρώπη θα σταματήσουν μέχρι το 2025. Όπως έχουμε την ιδιαίτερη αυτή περίπτωση Βουλγαρίας, Λιθουανίας και Σλοβακίας, βλέπουμε ότι ο αφοπλισμός αυτών των πυρηνικών αντιδραστήριων και η διαχείριση των αποβλήτων τους είναι κάτι που είναι τεχνολογικός περίπλοκο και είναι και μακρά διαδικασία και απαιτεί ουσιαστικούς οικονομικούς ε, πόρους για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την, την πυρηνική ασφάλεια στην Βουλγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία, οι χώρες αυτές δεσμεύτηκαν στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις να κλείσουν νωρί και να αφοπλίσουν οκτώ μη αναβαθμίσιμους πυρηνικού αντιδραστήρες, αναγνωρίζοντας τις εξαιρετικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες αυτών των δεσμεύσεών τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε οικονομική βοήθεια στις τρεις χώρες και στα προγράμματά τους έδωσε 2,8 δισεκατομμύριο ευρώ γενικά από το 1999 μέχρι το 2013. Βλέποντας πόσο σημαντικά είναι τα χρήματα αυτά, μεγάλο ποσό, και περίπλοκες απαιτήσει που υπάρχουν για τη διάλυση αυτών των αντιδραστήριων, ξεκίνησε το τρεχτικό συνέδριο τη εργασίας του τον Οκτώβριο του 2009. Η ειδική έκθεση εστιάστηκε στην εφαρμογή στο πρόγραμμα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω σε Βουλγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία από 99 μέχρι το τέλος του 2010 για την ε, διάλυση αυτών των αντιδραστήριων και εξετάσαμε κατά πόσο η δράση που η Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιστοιχούσαν στις ανάγκες κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν ως εσχεδιάστηκε και αν ήταν επαρκή τα κυβερνητικά μέτρα ούτως ώστε να είναι καλύτερη δυνατή χρήση των πόρων. Αυτός ο έλεγχος παρακολουθήθηκε με μεγάλο ενδιαφέρον και από πλευρά ελεγκτών, αλλά και από όλους τους ενδιαφερομένους. Προκατατικά πορίσματα του ελέγχου υποβλήθηκαν στην Επιτροπή σας και ο Μαρινέσκου συνέταξε ε, έκθεση γνώμη όσον αφορά τις πολιτικές συνέπειες και επιδράσεις αυτής της προσπάθειας. Στα πλαίσια συνεργασία ήταν καρποφόρες οι συζητήσεις που έγιναν με τον εισηγητή σα και το ελεκτικό συνέδριο ε, έδωσε στον κύριο Μαρινέσκου όλες σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται για να συνταχθεί το ψήφισμα της 5ης Απριλίου του 2011 της Επιτροπής όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης Ευρωπαϊκής Ενώσεως στον τομέα της, ε, του αφοπλισμού αυτών των πυρηνικών αντιδραστήρων στα κράτη-μέλη. Μετά από τα προκατατικά πορίσματα της εκθέσεώς μας, και σε αντίδραση αυτά και κατόπιν αναγνώσεω των συμπερασμάτων τη Επιτροπή σα, εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγηση συνεπιών και ένα νέο πλαίσιο διαδικαστικό που δημιουργήθηκε και που θέτει συγκεκριμένου στόχου, καθορίζει ρόλου, ευθύνε και απαιτήσει για εποπτεία και έλεγχο. Όλα αυτά καθορίζονται πολύ σαφέστερα μέχρι τώρα. Το ελεκτικό συνέδριο μετά την αντιφατική αυτή διαδικασία που ακολουθήθηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά αυτή την αντι... τη συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ολοκλήρωσε την έκθεση του το Φεβρουάριο του 2012. Αυτή η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ναι, μεν η Βουλγαρία, η Λιθουανία και η Σλοβακία έκλεισαν του αντιδραστήρε σύμφωνα με τι υποχρεώσει που είχαν αναλάβει και έχουν επιτευθεί τα σημαντικά, ε, οι σημαντικοί στόχοι όσον αφορά τον αφοπλισμό των αντιδραστήρων. Η βασική διαδικασία είναι ακόμα μπροστά μα και οι τελικές ε, φάσεις απαιτούν συμπροματική χρηματοδότηση, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σαν αποτέλεσμα του σχετικού, ε, σχετικά χαλαρού πλαισίου πολιτικής τα προγράμματα δεν έχουν υποστεί πλήρη εξολόγηση αναγκών, ε, θέση προτεραιοτήτων και συγκεκριμένους προς επίτευξη στόχους. Ο εντοπισμός των δραστηριοτήτων για τον αφοπλισμό των αντιδραστήρων εξακολουθεί. Μεγάλα προγράμματα υποδομών καθυστερούν και ξεπερνούν και τι προβλεπόμενε δαπάνε. Οι εκτιμήσει για τι δαπάνε δεν έχουν ολοκληρωθεί εν απουσία βασικών πληροφοριών όσον αφορά τα, α, τα ραδιενεργά απόβλητα και τις τεχνολογίες που απαιτούνται για την επεξεργασία των αποβλήτων. Μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων για να μειωθούν οι συνέπειες της πρώην, του πρώιμου κλεισίματος των πυρηνικών αντιδραστήριων είναι κάτι που χρηματοδοτήθηκε αλλά δεν ξέρουμε πόσο μειώθηκαν εντικές συνέπειες ε, και δεν είναι σαφείς οι ευθύνε. Δεν υπάρχει αξιολόγηση πλήρης ε, αναγκών, θέσεις προτεραιοτήτων και συγκεκριμένοι στόχοι. Η εποπτεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εστιάζεται επί της εκτελέσεως του προπολογισμού εν γέννη. Βάσει των πορισμάτων του, το ελεκτικό συνέδριο συνέστησε ότι πριν περαιτέρω δαπανηθούν χρήματα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλύσει τους διαθεσίμους πόρους και τα αναμενόμενα ωφέλη και να δημιουργήσει τις συνθήκες για αποτελεσματική, αποδοτική και οικονομική χρήση των πόρων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να καταρτήσει μια νεπτομερή αξιολόγηση αναγκών, εξετάζοντας την πρόοδο των προγραμμάτων μέχρι τώρα οι δραστηριότητες που απομένουν να γίνουν, να εφαρμοστούν και ένα γενικό σχέδιο χρηματοδοτήσεως θα πρέπει να εντοπίζει ε, τους πηγές για τη χρηματοδότηση. Αυτό με τη σειρά του θα πρέπει να οδηγήσει σε στόχους που θα χρηγραμμίζονται με τους πόρους και με δείκτες επιδόσεων οι οποίοι θα μπορούν ακολούθως να ελεγχθούν και να υποβληθούν ιδέες αναφορέ αν χρειαστεί. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει να δώσει περαιτέρω οικονομική βοήθεια για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αυτή η υποστήριξη θα πρέπει να εδράζεται επί αξιολογήσεως τη προστιθέμενη αξία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως μη της παρεμβάσεω, εντοπίζοντας τις βασικές δραστηριότητες αποπλισμού των αντιδραστήριων που θα χρηματοδοτούνται μέσω του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, λαμβάνοντα υπόψη και άλλε δυνατότητε χρηματοδοτήσεω όπω είναι τα διαθετικά ταμεία και εξασφαλίζοντας την τήρηση των επαρκών όρων για την εκταμείωση χρημάτων τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ε, μια σημαντική συνέπεια του ελέγχου μα ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή τη στην ειδική έκθεση συμφώνησε να εφαρμόσει τι συστάσει του ελεκτικού συνεδρίου μέσω των προτάσεών τη για βοήθεια τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω μετά το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχθηκε την ανάγκη που υπάρχει να διενεργηθεί μια αξιολόγηση αντικτύπου και να αναθεωρήσει του δείκτε επιδόσεων, ούτω ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν για την περίοδο που ακολουθεί το 2013, ακόμα και για αυτήν. Είμαι πεπισμένο ότι η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του Ελεκτικού Συνεδρίου και τη Επιτροπή σα μπορεί να δραματίσει σημαντικό ρόλο στην διαφύλαξη τη πρακτική εφαρμογή αυτών των σημαντικών δεσμεύσεων που ανελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βάσει τη εκθέσεω του Ελεκτικού Συνεδρίου και σε στενή συνεργασία μαζί μα, σε εκτελεστικό επίπεδο και στη δεύτερη έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου που αναλύει τον περίπλοκο χαρακτήρα των προγραμμάτων κλεισίματο αυτών των δραστήρων είναι ένα κείμενο που έχει συνταχθεί. Αυτό το σχέδιο κειμένου σωστά αναφέρεται σε αδυναμίε τη διαχειρίσεω των προγραμμάτων και την υλοποίηση αυτών. Τονίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν τα διάφορα χρηματοδοτικά κενά και υποστηρίζει την εξαίρεση περαιτέρω χρηματοδότηση μέτρων μετρίαση, επιμένει επί της ανάγκης διοργανώσεως του αφοπλισμού και κλεισίματος των αντιδραστήρων, τόσο ώστε να είναι κάτι αμετάκλητο, τονίζει την ανάγκη να πετευχθεί τεχνογνωσία που διαφέρει από τον τρόπο λειτουργίας του αντιδραστήρα, όταν μετακινείται από τη λειτουργία στην πάση λειτουργία. Τονίζει το έγγραφο την κρίσιμη σημασία που έχουν και η γενική και η λεπτομερή εκ των προτέρων αξιολόγηση, εντοπίζοντα τι ειδικέ δραστηριότητε που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν και την εφαρμογή των εκ των υστέρων συνθηκών πρέπει να επικρατούν σε σχέση με τους όρους που θα τίθεται για μελλοντικές εκταμίευσεις. Πέραν αυτών, η έκθεσή σας σωστά αναφέρεται στον προβληματικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας ανα, Ανεκοδομήσεως και Ανάπτυξης και την ανάγκη να υπάρχει καλύτερος μηχανισμός διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης και της εφαρμογής των σχετικών δικτών και θέτει ερωτήματα στον αφορά την προστιθέμενη αξία της μεταφοράς διαχειρήσεως προγραμμάτων σε αυτή την τράπεζα καλεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεων Ενικοδομήσεω να διαθέσει στο Κοινοβούλιο τι σχετικέ εκθέσει όσον αφορά την εφαρμογή των ε, μέτρων και των έργων και ζητά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την προστιθέμενη αξία τη συνεργασία με την Λόγο Τράπεζα. Εμείς από την πλευρά μας ελπίζουμε ότι αυτές οι δικαιολογημένε ερωτήσεις θα απαντηθούν σωστά και προσφέρουμε σε εσά τη βοήθειά μας και τη συνεργασία μας επί τη βάση της εμπειρίας μας και τη θεσμική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Νοικοδόμησης και Ανάπτυξη, ούτω ώστε να καταλήξουν σωστή αξιολόγηση και επίλυση του προβλήματο. Ελπίζω ότι οι εκθέσεις του Δικαστηρίου και τη Επιτροπή σα μπορούν να παράσχουν σημαντική βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προετοιμάσει εκείνοι βιώσιμε προτάσει που θα βοηθήσουν του λαμβάνοντα την απόφαση να αξιολογήσουν την προστιθέμενη χρηματοδότηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση που απαιτείται, τόσο ώστε με ασφάλεια να εφαρμοστούν ε, τα προγράμματα και διαδικασία αφοπλισμού των αντιδραστήριων η πρακτική εφαρμογή των προτάσεων που θα ακολουθήσει θα πρέπει να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των προγραμμάτων αφοπλισμού στη Βουλγαρία, Λιθουανία και Σλοβακία, αυξάνοντα την πυρηνική ασφάλεια σε όλη την Ευρώπη του τρόπο και συμβάλλοντα στη βελτίωση της ζωή, τη ποιότητα ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Κυρία Πρόεδρε, δράτω με τι ευκαιρίε να σα διαβεβαιώσω και εσά και το να σας πω ότι το συνέδριο έχει δεσμευτεί να συνεργάζεται στενά με τον εισηγητή σας, τον κύριο Μαρινέσκου και με όλους σας, αξιότιμα μέλη αυτής της Επιτροπής, τόσο ώστε να διευκολυνθεί η προετοιμασία, η υιοθέτηση και εκτέλεση των σημαντικών αυτών βημάτων και μέτρων που αναφέρονται και στις δύο εκθέσεις μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση. Ο κύριος Μαρινέσκο, ηγητής μας, θα πάρει το λόγο τώρα. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση του ελεκτικού συνεδρίου. Σας ευχαριστώ και τα μέλη μου του ελεκτικού συνεδρίου, με τα οποία υπήρξε άριστη συνεργασία. Ναι, ήδη στην πρώτη έκθεση για το ίδιο θέμα θα θέσει στη διάθεσή μου πάρα πολλές πληροφορίες και το πράξετε και αυτή τη φορά και σας ευχαριστώ πολύ. Ε, παράλληλα με την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου διάβασα την πρώτη έκθεση την οποία ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ανέλησα. Και αυτό ισχύει και το διάστημα από το 14 έως το και για τα ποσά τα οποία χορηγήθηκαν για τον παραπλησμό των πυρηνικών σταθμών. Πρόκειται για κάποιους πυρηνικούς αντιδραστήρες ε, στις ε, τρεις αυτές χώρες που συζητούμε εδώ. Βεβαίως είμαι ανοιχτός και θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη των συναδέλφων και η έκθεσή μου είχε κυρίως σαν στόχο το να τονίσει τα εξής θέματα. Πρώτον, χρειάζεται ε, ιδιαιτέρως ε, αυστηρός προγραμματισμός με αυστηρή τήρηση των προθεσμιών. Και θα πρέπει να σκεφτούμε σε σχέση με έναν προϋπολογισμό και να δούμε πώς μπορεί να χρηματοδοτηθεί κάθε δραστηριότητα. Και βεβαίως θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης. Αυτά τα δύο στοιχεία θα πρέπει να αποτελούν προϋποθέσεις για την εκταμιεύση των ποσών ε, και για την έγκρισή τους μέσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και αυτό γιατί θα πρέπει να το κάνουμε για το χρονικό διάστημα από το 14 στο 20, δηλαδή την διανομή αυτών των κονδυλίων. Και στη συνέχεια θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα ποσά αυτά θα εξυπηρετήσουν μόνο το σκοπό του παροπλισμού των πυρηνικών σταθμών και δεν θα διοχετευτούν σε άλλες ε, ε, δραστηριότητες και θα πρέπει οπωσδήποτε να διευκρινίσουμε κατά πόσο αυτά θα είναι τα τελευταία χρήματα τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει των συνθηκών θα, ε, θα δώσει για αυτές τις ε, δραστηριότητες του παροπλισμού. Και θα πρέπει επίσης να διευκρινίσουμε κατά πόσο αυτή η συνεργασία εξακολουθεί να είναι αναγκαία γιατί οι σημαντικές ε, πηγές χρηματοδότησης μέχρι στιγμής ε, πηγάζουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο χρειαζόμαστε άλλες πηγές χρηματοδότησης. Τα χρήματα τα οποία δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ε, θα δώσει μάλλον για την περίοδο αυτή 14 έως 20 θα πρέπει να ελεγχθούν ε, αυστηρά και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στον ε, κανονισμό και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα πρέπει να έχει μόνον το ελεκτικό συνέδριο τον ε, έλεγχο για αυτά τα κονδύλια. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της έκθεσής μου και βεβαίως βρίσκομαι στη διάθεσή σας για να προχωρήσουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων. Περιμένω τα σχόλιά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Παρινέσκου. Τώρα η Επιτροπή που αντιπροσωπεύεται από τον Πίτερ Φάρας που είναι ε, στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Φαζάκας για την παρουσίαση της έκθεσης. Εάν ανατρέξουμε στο ιστορικό κομμάτι θα διαπιστώσουμε ότι η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου είναι καλά ισορροπημένη. Τα σχόλια της έκθεσης για αυτή την έκθεση έχουν δημοσιοποιηθεί Άρα λοιπόν θα ήθελα να επικεντρώσω την προσοχή μου στην ε, έκθεση του εισηγητού του κυρίου Μαρινέσκου, τον οποίον θέλω να ευχαριστήσω με την ευκαιρία αυτή για την παρουσίαση αυτού του σχεδίου έκθεσης. Εν γέννη πιστεύω ότι η Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως τα συμπεράσματα του σχεδίου έκθεσης έτσι όπως παρουσιάστηκαν από τον κύριο Φαζάσκας και αυτά τα συμπεράσματα κατά κάποιο τρόπο επικαλύπτονται από την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση από το 2014 έως το 2020. Και υπογραμμίζεται ότι η οικονομική ευθύνη για, την, για τον παροπλισμό εναπόκειται στις χώρες μέλη και εμείς δεν μπορούμε παρά να προσυπογράψουμε αυτή τη βασική αρχή. Επίσης συμφωνούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ένα ξεκάθαρο ε, σχέδιο χρηματοδότησης ε, και θα πρέπει να ανοιχνευτούν οι πηγές ε, χρηματοδότησης. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να δείστε κατανόηση του το γεγονός ότι δεν μπορεί η Επιτροπή να το πράξει αυτό από μόνη της. Ε, γιατί δεν έχουμε πρόσβαση στα εθνικά κονδύλια που είναι διαθέσιμα και, για την, ε, και στην ε, ανάπτυξη αυτών των κονδυλίων. Και εφόσον επόκειται στην εθνική αρμοδιότητα θα πρέπει τα εθνικά αυτά κονδύλια να συμπεριληφθούν στα προγράμματα. Επίσης έχουμε προτείνει και δηλώσει ότι η οικονομική συνδρομή της Ευρωπαϊκής θα πρέπει να συνεχίσει μετά το 2020 και θα πρέπει να υπάρξει μια αυστηρή ε, παρακολούθηση και θα πρέπει να διατυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι όροι όπως και να συμπεριλαμβάνονται στην ε, πρωταθήσα νομοθεσία και θα πρέπει αυτό να αρκεί. Μαζί με τον εισηγητή έχουμε επίσης την άποψη ότι κάποια μέτρα μετρίασης δεν θα πρέπει πλέον να εφαρμόζονται μετά ε, το, την κάλυψη κάποιων ελλείψεων και χασμάτων όσον αφορά τον παραπλησμό γιατί οι απαιτήσει αυτές έχουν ε, πληρωθεί. Όπως ε, ε, καλεί τόσο το ελεγκτικό συνέδριο όσο και ο εισηγητής, Βεβαίω θα κάνουμε μια αξιολόγηση εν σχέση με την καλύτερη δυνατή χρηματοδότηση και υποστήριξη αυτών των σχεδίων στον μέλλον και έχουν ε, γίνει αναφορές στη μελλοντική μας συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση. Και εμείς στη δική μου διεύθυνση θα, κάνουμε, θα προβούμε σε μια ανάλυση της κατάστασης. Κύριε Πρόεδρε, ε, θα θέλαμε να πούμε ότι χαιρετίζουμε κατακλείδη το έργο του εισηγητού και υποστηρίζουμε όλα τα συμπεράσματα. Υπάρχουν βεβαίως κάποια ε, σημεία όπου θα ήμουν διατεθειμένος να θέσω στη διάθεση του εισηγητού κάποια κείμενα γιατί βρισκόμαστε σε ένα κόσμο εξελίξη και οι δύο αναφέρθηκαν σε, στα 143 πυρηνικούς σταθμούς που λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις γιατί μετά το ατύχημα της Φοκουσίμα οι Γερμανοί έκλεισαν πολλούς πυρηνικούς σταθμούς που λειτουργούσαν πριν από τη Φοκουσίμα, αλλά νομίζω ότι μπορούν ε, να γίνουν αυτές οι διορθώσεις ε, συνεργασία με τον εισηγητή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Φάρας. Ε, συνάδελφοι, εάν θέλετε, έχετε το λόγο. κύριος Μπαλσίτης θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ. Πράγματι, ο παροπλισμός του πυρηνικού, των πυρηνικών σταθμών ήταν βασικό θέμα σε μια έκτακτη συνεδρίαση η οποία έγινε την περασμένη, έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα και θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τον συνάδελφο κύριο Μαρινέσκου για την έκθεσή του και θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι για το γεγονός ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ιδιαίτερως ακριβείς και ευσταθούν. Έχω κάποιες ανησυχίες όσον αφορά τα όσα είπε εκπρόσωπος της Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να είναι αρμόδια για, την, για τον οριστικό παροπλισμό αυτών των πυρηνικών ε, σταθμών. Ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να τηρήσουμε τις βασικές ε, αρχές. Ε, τη συνθήκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός ο οποίος ε, παρέχει τη χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι και αρμόδιος για την χρήση αυτών των κονδυλίων. Και κατ' ουσία βρισκόμαστε ενώπιον αυτού του προβλήματος. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης, η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία παροπλισμού ιδιαιτέρως του πυρηνικού σταθμού της Ιγναλίνα της Λιθουανίας. Η τράπεζα αυτή καθόρισε το πώς ε, θα πρέπει να υπογραφούν οι δημόσιες συμβάσεις και σε ποια χρονικά διαστήματα θα πρέπει να επιληθούν ποια προβλήματα. Τώρα όσον αφορά αυτό όσον αφορά το ιστορικό. Αλλά βεβαίω δεν πρόκειται για ένα κυρίω οικονομικό ζήτημα, αλλά πρωτίστω πολιτικό. Κάτι τη διάρκεια της προσχώρησή μας το έτος 2004 η, η δική μας για την ενέργεια δεν έγιναν καλώς ε, κατανοητοί στη Λιθουανία. Δεν ακούστηκε η φωνή τους. Και ε, παρόλο που ε, διατυπώθηκε ο ισχυρισμό ότι το, και διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι το πυρηνικό σταθμό ε, τη Σιγναλίνα μπορεί να λειτουργεί χωρί προβλήματα μέχρι το 2017. Αυτό τη ισχυρίστηκε η κυβέρνηση. Ωστόσο, είχαμε υπογράψει ένα πρωτόκολλο το οποίο προέβλεπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χορηγήσει μια οικονομική συνδρομή, ούτω ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί ο παραπλησμό του πυρηνικού σταθμού. Βεβαίω, η χρηματοδότηση δεν ήταν υπαρκή και μέχρι το 2014 δεν ε, ήταν αρκετά τα κονδύλια αυτά, αλλά τώρα έχουμε αναλάβει αυτή την πολιτική δέσμευση και ε, βεβαίως κατανοούμε το ότι το 2020 ε, θα σταματήσει η οικονομική ε, συνδρομή αλλά είναι πιθανό μέχρι τότε μέχρι το 2020 να μην έχει ολοκληρωθεί ο παραπληκτισμός και τότε θα τεθεί το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας ε, και θα πρέπει εν πάση περιπτώσει να αποφύγουμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση. Ε, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα πρέπει και η Κομισιόν να εκπληρώσει το δικό της ρόλο όσον αφορά ιδιαιτέρως τις ε, αρμοδιότητες όλων των ενεχόμενων ε, μερών. Και εγώ θεωρώ ότι ένα οριστικό παροπλισμό θα πρέπει να παραμείνει αρμόδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να διατυπώσει συγκεκριμένου στόχου, θα πρέπει να θέσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, να ονομάσει συγκεκριμένε ημερομηνίε και να καταρτήσει ε, προγράμματα ελέγχου και βεβαίως οι εκθέσεις αυτές θα πρέπει να μπορούν να συζητώνται σε διάφορα επίπεδα, ιδιαίτερως στο επίπεδο που ε, διαπιστώνονται κάποιες ε, ελλείψεις. Είμαι πεπισμένος ότι με τις προσπάθειες της Επιτροπής ε, Προπολογισμών και με τις προσπάθειες της Επιτροπής θα μπορέσουμε να εκπληρώσουμε αυτές τις υποχρεώσεις. Η κυρία Γκρέσλε έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όλη αυτή όλη η έκθεση με αφήνει άφωνη. Δώσαμε 2,8 δις ε, και λέει το ελεγκτικό συνέδριο ότι θα χρειαστούν άλλα 2,8 δις και παρόλα αυτά δεν είναι αναστρέψιμος ε, ε, δεν είναι μη αναστρέψιμος μάλλον ο παραπλησμός των πυρηνικών σταθμών. Το ερώτημά μου είναι τι καταφέραμε με αυτά τα 2,8 δις. Είναι φυσιολογικό κάτι τέτοιο. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Ε, τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες. Τι γνωρίζουμε όσον αφορά τις προκηρύξεις διαγωνισμών. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θεωρώ ότι δεν έχει απαντηθεί επαρκώ. Θεωρώ ότι η έκθεση είναι μεν ενδιαφέρουσα, αλλά θα μπορούσε κατά την άποψή μου να είναι πιο λεπτομερής, πιο μακροτενή. Ε, και υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία στα οποία θα έπρεπε να εμβαθύνουμε. Τον Ιούλιο θα πάμε στην Λιθουανία, στην Ιγκναλίνα συγκεκριμένα και το δεύτερο ερώτημά μου εδώ είναι ποια είναι τα ερωτήματα που θα έπρεπε να θέσουμε. Δηλαδή τι σκέφτεστε ότι θα πρέπει να θέσουμε ως πρόβλημα. Ποια είναι τα σημεία που θα πρέπει να επεξεργαστούμε τώρα σαν αφορά την εξέλιξη του κόστους. Και θα ήθελα επίσης να πω σαν εισηγή το Μάριαν, στην πρώτη σου έκθεση, στην έκθεση πρωτοβουλίας, ε, αναφέρει σε μια ετήσια έκθεση της Κομισιόν όσον αφορά τις ε, πρόοδους. Ζήτησε μια τέτοια έκθεση, η οποία πλέον όμω δεν αναφέρεται εδώ και δεν συμπεριλαμβάνεται. Και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθεί μια τέτοια έκθεση της Επιτροπής. Τώρα, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, θεωρώ ότι υπάρχει κάποια οριστία στην έκθεση. Δεν παίρνει τελικά θέση. Και μπορώ να καταλάβω βεβαίω ότι κρεμεί το θέμα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με αυτά τα ερήπια τα οποία ε, συνεχίζουν να υπάρχουν και όπου υπάρχει τεράστια αοριστία και ασάφεια με το πώς θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Ο κύριος Μόλτερ έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ. Διάβασα την έκθεση, Πρόεδρε, και το γενικό παράπονο, αν θέλετε, είναι ότι δεν είναι επαρκής ε, ο σχεδιασμός, ε, δεν υπήρχε εξάντα κτλ. Αλλά ένα από τα βασικά σημεία, κατά τη γνώμη μου, είναι στο 2, εκεί που μου μιλάει για την θεωρητική ημερομηνία παύση και αναφέρεται ένα αριθμό ετών, ε, σε τις περιπτώσεις όμως έχουμε υπερβεί αυτή την πρόβλεψη. Ε, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν υπήρξε επαρκής πρώτερος σχεδιασμός. Ε, θα πρέπει να κλείσουν το νωρίτερο δυνατό αυτή η πυρηνική σταθμή. Για την Ιγναλίνα λέτε παραδείγματος χάρη ότι η μονάδα 1 ε, θα πρέπει να κλείσει το 2013. Μα αφού είχε κλείσει ήδη το 2004 και πιστεύω ότι αυτό είναι θετικό σημάδι για το μέλλον. Θα ρωτήσω λοιπόν, από όσα καταλαβαίνω, ότι παρά το σχεδιασμό, παρά την εξαναταξιολόγηση και παρότι είναι ορθή χρήση των ε, κονδυλίων, τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον από την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείτε ότι υπάρχει το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο βάση και της έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου. Από ό,τι θυμάμαι για την ε, στη Λιθουανία ένα μεγάλο κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας ε, παραγόταν από αυτό το σταθμό. Ποια είναι λοιπόν η αναλλακτική πηγή. Η Λιθουανία έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με το ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει βρεθεί λύση και πρέπει να συνδράμουμε και για αυτή τη λύση. Ευχαριστούμε κύριο Γκάγια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι... Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συζητήσουμε για δύο μεγάλα προβλήματα και να δούμε ε, το εξή. Στην ψηφορία για την έκθεση αυτή θα πρέπει να ασχοληθούμε ξεκάθαρα με αυτά τα προβλήματα. Ε, πριν από λίγο καιρό, στα πλαίσια της κατάρτισης του προπολογισμού, είχαμε μία μακρά συζήτηση με το Συμβούλιο εν σχέση με το πώς η εξέλιξη του κόστος για τον παραπληπισμό των τριών πυρηνικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να παρουσιαστεί. Και όταν ακούσω εδώ τι γίνεται με το με δημοσιονομικό πλαίσιο, θεωρώ ότι οδηγούμεθα σε ένα αδιέξοδο. Και αν δούμε τι γίνεται με τις διάφορες χώρες μέλη όπου λένε ότι θέλουν να μειώσουν τον προπολογισμό και όπου εμείς από την άλλη ταυτόχρονα λέμε ότι όσον αφορά την εξέλιξη του κόσμου για τον παραπληκτισμό των τριών πυρηνικών σταθμών θα ανακύψουν ε, περαιτέρω έξοδα ε, βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θα πρέπει πραγματικά να συζητήσουμε λεπτομεριακά ποιες είναι οι ιδέες που έχει το Κοινοβούλιο όσον αφορά τις δαπάνες αυτές που πρόκειται να προκύψουν. Ε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να συμμετάσχει όλο το Κοινοβούλιο και όχι μόνο η Επιτροπή αυτή σε σχέση με το ζήτημα αυτό επιπλέον, των επιπλέον δαπανών. Τώρα, έχω μία ερώτηση για το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή. Κατά πόσο γνωρίζουμε ακριβώ, κατά πόσο τα κονδύλια τα οποία δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στι χώρε μέλη για τον παραπλουσμό των πυρηνικών σταθμών, πώ χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα κονδύλια. Και τα λέω αυτά με το εξή σκεπτικό ε, μια γερμανική εταιρεία συμμετείχε σε ένα από αυτά τα προγράμματα παροπλισμού και είχε κάποιες ε, δυσκολίες πληρωμής γιατί τελικά δεν ε, πληρώθηκαν τα χρήματα ε, στους δικαιούχους. Και από τη μία λοιπόν διαπιστώνουμε ότι δίδονται χρήματα αλλά τελικά οι χώρες μέλη δεν κάνουν καθαρό παιχνίδι, δεν τηρούν το χρονοδιάγραμμα και από την άλλη οι εταιρείε που συμμετέχουν τελικά περιμένουν να καλυφθούν τα έξοδά τους. Και ε, ρωτώ πού βρίσκω, πού πήγαν αυτά τα κονδύλια. Και θα ήθελα να προτιμάσω ορισμένες τροπολογίες για να συμπεριληφθούν ενδεχομένω στην έκθεση του κυρίου Μαρινέσκου. Και θα ήθελα εγώ από αυτό το βήμα να θέσω ξεκάθαρα το ερώτημα. Τι γνωρίζετε επακριβώς για το πώς χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε. Εφόσον πολλές ερωτήσεις απευθύνονται προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ζητήσω πρώτα απ' όλα από το Ελεγκτικό Συνέδριο να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τι ευχαριστίες μου προ την Επιτροπή Ελέγχου των Προπολογισμών και όλα τα μέλη τη για το ενδιαφέρον που δείχνουν για αυτό το καυτό, θα τολμούσα να το αποκαλέσω ζήτημα, που είναι τόσο σημαντικό για όλου μα. Ήμουν και εγώ μέλος της Επιτροπής σας και χαίρομαι που ανέλαβα τον έλεγχο από πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου, διότι θυμάμαι ότι και νωρίτερα από το 2004 όταν ήμουν ακόμη εδώ, αυτό το θέμα ετίθετο με τον εξή τρόπο. Με, για ποιο λόγο δαπανά τόσα χρήματα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ποιο είναι το απτό αποτέλεσμα τη χρήση του. Θα έλεγα λοιπόν πρώτα απ' όλα, με την ιδιότητα που έχω τώρα του μέλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ε, είναι επαγγελματικό καθήκον του ελεγκτικού συνεδρίου να δώσει στην αρχή χορήγηση απαλλαγή σε καλά ε, τεκμηριωμένες αποδείξεις ε, μετά από τη διεξαγωγή του ελέγχου. Κατόπιν ε, η δική σας επιτροπή, οι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν την ευθύνη βάσει αυτών των στοιχείων να λάβουν και τις σωστέ αποφάσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι κυρίω πολιτικέ οι αποφάσεις και το ελεγκτικό συνέδριο είναι στην η υπηρεσία σας, αλλά δεν θα καταλήξουμε εμείς στη θέση σε συμπεράσματα. Θα αρχίσω τώρα από τα σχόλια του κυρίου Μπαλσίτη, δεν ξέρω αν προφέρω και σωστά το όνομά του λέγοντας ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά ιδιάζουσα περίπτωση. Θα θυμάστε ίσως σε μια σύσκεψη διαπραγματεύσεων με όλες τις νέες χώρες και τη δική μου, την Ουγγαρία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε πάυση ή λειτουργία ε, των υφιστάμενων πυρηνικών σταθμών. Στην περίπτωση τη Ουγγαρία, ε, η λειτουργια των εφισταμενων πυρηνικων σταθμων στην περιπτωση τη ουγγαρια η χωρα μου κατάφερε να εξηγήσει και να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όλοι οι πυρηνικοί μας σταθμοί συνάδουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στην περίπτωση της Λιθουανίας, όπως είπε ο κ. Βελτέσης, δεν ε, ήταν πολύ δυσαρέστη έκπληξη όταν ε, έλαβαν ε, το αίτημα του κυρίου Φερχόγγεν ότι πρέπει να προβείτε στην πάυση νωρίτερα από ό,τι το προβλεπόμενο. Στη συνέχεια υπήρξε μια συμφωνία που προέβλεπε το πολύ σημαντικό αντίκτυπο από οικονομικής και κοινωνικής πλευράς της πάυσης λειτουργίας, εξού και η ιδέα να συνδράμει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κόστος. Ελέγξαμε αυτή τη συμφωνία και συνειδητοποιήσαμε ότι είναι πάρα πολύ ανοιχτή. Δηλαδή το πλαίσιο δεν σα δίνει ούτε το ποσό, ούτε τις, ε, το, τους τίτλους τα κεφάλαια. Υπάρχει μόνο μία ανάληψη υποχρέωση από της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα συμβάλλει στις ε, δαπάνες. Ε, αυτό όμως είναι μια αντίφαση και στρέφομαι προς τον συνάδελφο για να διαφωνήσω. Ζητώ συγγνώμη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να καταβάλει το κόστος του παροπλισμού. Διότι αν αντελήθην ορθά ε, την γνωμοδότηση του της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη θέση του Κοινοβουλίου, ακολουθούμε την αρχή ο πληρώνει και άρα η χώρα πρέπει να καταβάλει το κόστος και ε, καθήκον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να σας ε, βοηθήσει ούτως ώστε να συμμορφωθείτε με όλα αυτά τα κριτήρια. Σε απάντηση στην έκθεσή μα, απάντησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ερμηνεύουν αυτή τη συμφωνία ω πράξη αλληλεγγύη. Πολύ ωραία ακούγεται από πολιτική άποψη, αλλά κανεί δεν ξέρει τι εννοείται. Τι εννοείται λέγοντα πράξη αλληλεγγύη, Αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου το κόστο του παροπλισμού. Τι εννοείται με την αρχή τη ε, mitigation, μέχρι πού μπορείτε να καλύψετε το κόστο τη άμβληση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών και απαντώντα τώρα στην αξιότιμη συνάδελφο κυρία Γκρέσλε θα της πω ότι σε όλους τους ελέγχους ε, λειτουργήσαμε εξονυχιστικά και όπως είπε και ο κύριος Μόλτερ διαπιστώσαμε ότι ήταν ε, ε, ορθή η εκταμίευση, η χρήση των κονδυλίων δεν σημειώθηκε καμία παρατυπία σε σχέση με την βάση λειτουργία, τον παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών και την άμβλυνση των οικονομικοκοινωνικών συνεπειών. Ε, και ήταν και κινούμενο ο στόχο, και όχι μόνο κινούμενο, ήταν και αόρατο, διότι πριν από 10 χρόνια κανεί δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσει πώ ενδεχομένω θα κόστιζε ένα παροπλισμό. Ε, ζητώ συγγνώμη που το λέω, αλλά χαίρονταν που γινόντουσαν βήματα, αλλά στόχο δεν υπήρχε. Πραγματική αξιολόγηση δεν υπήρχε. Τι εννοείται με ε, τον πυρηνικό παροπλισμό, τι ενδέχεται να κοστίσει και ούτω καθεξής. Τότε λοιπόν ήταν όλοι ευχαριστημένοι και σας έλεγαν όλοι ότι η χρήση των κονδυλίων δεν σημειώνει καμία παρατυπία. Για να απαντήσω στην κυρία Γκρέσλε θα πω τα εξής. Ε, κάλυψαν αυτή την υποχρέωση που είχαν αναλάβει. Έχουν κλείσει οι πυρηνικοί στοθμοί. Βέβαια, σωστά λέει ο εισηγητή σα ε, και επικρίνει, διότι δεν μπορεί να θεωρήσει κανεί ότι είναι μια αναστρέψιμη μια πάυση λειτουργία. Θα ήθελα να σα παραπέμψω σε διάφορε ε, ε, εξαγγελίες ε, από πλευράς της Βουλγαρίας το 2009 θα θυμάστε ότι υπήρχε έλλειψη ως προς τροφοδότηση σε φυσικό αέριο και πρότεινε η Βουλγαρία μελητή και λόγω της κρίσης ε, στην τροφοδότηση σε αέριο ζήτησε λοιπόν μία εξαίρεση να επαναλειτουργίας του Κοσλοντούι και έχω μαζί μου τα σχετικά έγγραφα στη Λιθουανία πριν από τρεις μήνες τώρα ε, υπήρξε ένα δημοσίευμα του τύπου βάσει του οποίου αν η Λιθουανία δεν λάμβανε αρκετά κονδύλια από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επανεξέτασε το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας των πυρηνικών σταθμών. Το κόστος καλύφθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν για την πάυση λειτουργίας. Δυστυχώς όμως η διαδικασία δεν μπορεί να θεωρηθεί μη αναστρέψιμη διότι ο παρεπλισμός ε, επί της δεν συνέβη ποτέ για να είμαστε σίγουροι ότι είναι ε, η χρήση των κονδυλίων ε, για να βγει ένα συμπέρασμα. Καταλαβαίνετε, δεν μπορείτε να βασιστείτε στη δική μας την απόφαση του ελεγκτικού συνεδρίου. Εμεί ελέγχουμε. Εσείς θα αποφασίσετε, εσείς στο πολιτικό όργανο, αν στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό θα πρέπει να προβλέψετε και άλλα ε, κονδύλια. Επιλύσατε για 550 εκατομμύρια αλλά δεν φτάνουν αυτά τα χρήματα. Ούτε πολύ λίγα είναι, ούτε πάρα πολλά και δεν μας φτάνουν. Επίσης χρειάζεται και η εξάντη αξιολόγηση. Να ξέρουμε κάθε πρόγραμμα τι θα κοστίσει και πρώτου εκταμιεύσουμε, αντί για 2,5 εκατομμύρια θα περάσουμε στα 550, να γνωρίζετε ότι θα πρέπει να αιτιολογηθούν τα επιπρόσθετα κονδύλια με αυτόν τον τρόπο. Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναρωτηθείτε τι έκανε με αυτό το κινούμενο στόχο. Έδωσε τη διαχείριση στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, ε μα είναι τράπεζα όμως. Όταν έχει τράπεζα, ε, ε, η τράπεζα λεφτά, δίνει ε, λεφτά, αλλά δεν ελέγχει τη χρήση τους. Δική σας δουλειά είναι να ελέγξετε πώς ήταν η χρήση του και εμείς βάσει της δική μας έκθεση μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν σημειώθηκε παρατύπια, δεν σημειώθηκε απάτη. Οπότε δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε το πόρισμα τη προηγούμενη έκθεση να στραφείτε δηλαδή προ τον Όλφ. Όμω κατακρίνουμε ε, την προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Νοικοδόμηση, ε, η BRD, για αυτό το ρόλο. Σίγουρα τα χρήματα πήγανε σε ένα ε, διεθνές ταμείο παροπλισμών, αλλά οι υπόλοιποι δωρητές δεν συνέβαλαν τελικά. Και το θέμα είναι ο στόχος. Ε, θέλουμε να είναι μη αναστρέψιμη η υπάρξη λειτουργίας, ναι ή όχι. Αυτές είναι οι βασικές απαντήσεις που θα δώσω σε ερωτήσεις σας. Τώρα σε σχέση με αυτό που ρώτησε η κυρία Ίγκεμπορ Γκρέσλε. Τι θα συστήνατε εσείς στη Λιθουανία. Πρώτον, ε, να ε, διαπιστώσετε σε ποιο βαθμό είναι πραγματική η δεσμευσή τους. Κατανοούν ότι πρέπει να κλείσουν οι πυρηνικοί σταθμοί της Ιγναλίνα και ότι πρέπει να παροπλιστούν, διότι αυτό είχαμε συμφωνήσει στο παρελθόν. Πρέπει να καταλάβουν επίσης ότι δεν πρέπει να ε, χρησιμοποιούν, να εκμεταλλεύονται την τωρινή κατάσταση για να ε, επιστρέψουν σε διαπραγματεύσεις. Ε, το ελεγκτικό συνέδριο σωστά λέει στην έκθεση του ότι πάνω από 80% των κονδυλίων διοχετεύθηκαν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Στην περίπτωση της Λιθουανίας και κατόπιν αιτήματο της χώρας δημιουργήθηκε και ένας παράλληλος διάβλος ε, και εγώ αναρωτιέμαι γιατί χρειαζόταν, γιατί είμαι ειδικό σε αυτά τα θέματα, γιατί παράλληλος διάβλος, γιατί έγινε αξιολόγηση αντικτύπου. Ε, ε, όταν ε, διοχετεύτηκαν τα κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Νοικοδόμησης ε, και στην περίπτωση της Λιθουανίας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ένα άλλο κριτήριο. Ποιο είδους προσθέμενη αξία επιδιώκουμε με αυτήν την ειδική για τη Λιθουανία λύση είναι κέριο το ζήτημα όπως επίσης και αυτό της mitigation, της άμβλησης των οικονομικοινωνικών συνεπειών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, αλλά έχουν λάβει ε, στήριξη από τα διαρθρωτικά ταμεία όλες αυτές ε, οι χώρες. Αυτά τα κονδύλια πρέπει να χρησιμοποιήσουν για αυτό το σκοπό. Τα υπόλοιπα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τον παροπλισμό υπό την προϋπόθεση ότι χορηγείται εξάνταξιολόγηση και ότι οι δαπάνες ε, ε, γίνονται με ορθό τρόπο και προσφέρουν κυρίως ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Φάρας, τώρα θα θέλατε κι εσείς να προσθέσετε κάποια σύντομα σχόλια. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα όσον αφορά το ιστορικό και μετά θα μπω στα ερωτήματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα λειτουργούσε εντός του δέοντος νομικού πλαισίου. Αυτό προλεπόταν από τις ε, συνθήκες προσχώρησης. Υιοθετήθηκαν αυτές από όλα τα κράτη-μέλη. Και βασικό στόχο έθεσαν το ταχύ κλείσιμο των αντιδραστήρων που θεωρούνται οικονομικώς μη αναβαθμίσιμοι. Γι' αυτό δεν ανελήφθη μακρύ τέλειο σχεδιασμό όσον αφορά τον παροπλισμό των αντιδραστήρων. Αυτά πρέπει να τα δούμε διότι έγιναν κατά μία περίοδο ήταν πολύ κοντά χρονικά στη, στο ατύχημα του Τσέρνομπιλ. Για τις συγκεκριμένες ε, ερωτήσεις που ετέθησαν, κατά πόσο ε, είναι αμετάκλητο γεγονός το κλείσιμο των ε, αντιδραστήρων. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό δεν είναι δεδομένο όπως το Ιγναλίνα, στον αντιδραστήρα 2 της Ιγναλίνα. Γιατί? Διότι ο πυρήνας του αντιδραστήρα δεν μπορεί να εκενωθεί Διότι τα καύσιμα, ε, η ράβδη των καυσίμων είναι πλήρης, η χώρη των καυσίμων είναι πλήρης ε, και δεν έχει ολοκληρωθεί εκένωση. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην Πουχουνίτσα 1 και 2, Ήδη έχουν δοθεί άδειε παροπλισμού. Δεν λειτουργούν ε, πλέον εκεί ε, αυτοί οι αντιδραστήρες, αυτού ο αντιδραστήρες, αυτή η μονάδα. Και ποια ήταν η εναλλακτική λύση όσον αφορά το πρώιμο κλείσιμο. Η Ιγναλίνα, ο αντιδραστής Ιγναλίνα ήταν ο μεγαλύτερος αντιδραστήρας στην ιστορία. 70% της ηλεκτρικής ενέργειας της Λιθουανίας παρήχε μέχρι τότε. Και ήταν σημαντικότατο να ληφθούν μέτρα μείωση των συνέπειων. Διότι από τη μία μέρα στην άλλη έκλεισε το 35% τη μία μέρα και το 35% της παραγωγής την άλλη μέρα. Τι έκανε σαν αυτά τα μέτρα μειώσεως των αποτελεσμάτων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναβαθμίσαμε θερμικές μονάδες για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάντα μέσα στα περιβαλλοντικά πλαίσια και προδιαγραφές. Και ολοκληρώνεται και η κατασκευή μιας άλλης εγκαταστάσεως παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο. Είναι γνωστό το πώς ξοδεύτηκαν τα χρήματα, κυρία Πρόεδρε δεν υπήρξαν περιπτώσεις απάτης όπως αναφέρθηκε. Και πέρα από τον έλεγχο του ελεκτικού συνεδρίου, για φέτος έχουμε αναθέσει δύο λεπτομερείς ελέγχους, όπως κάναμε για Μποχουνίτσα, για Κοσλοντούι και, και για την Ιγναλίνα. Και στην περίπτωση του αντιδραστήρα της Ιγναλίνα δεν κρύψαμε ποτέ ότι υπάρχουν ε, καθυστερήσεις και εμπορικές διαφορές μεταξύ συμβαλωμένων μερών και εργοδοτών. Το αξιότιμο μέλος θα αναφερόταν, πιστεύω, σε συγκεκριμένη περίπτωση όπου κάποιο συμβαλόμενο μέρος, κάποιος ανάδοχος, ήδη κατασκεύασε ε, το χώρο για την το, το σκέπαστρο για την προσωρινή αποθήκευση των καυσίμων, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή, διότι υπάρχει εμπορική διαφορά κατά πόσο αυτά τα καλύματα που δόθηκαν επί τόπου παραδόθηκαν ε, εκτελούν το σκοπό τους. Είναι γνωστά αυτά, ασχολούμαστε με αυτά. Σε επίπεδο σχεδίων απορρίπτουμε αυτό που είναι σωστό. Προσπαθούμε να, να οι διαφορές και να καταβληθούν τα τελικά ποσά, να μην υπάρχουν καθυστερήσεις διότι υπάρχουν τα χρήματα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Φάρος. Κυρία Ρέστη. Ε, θα ήθελα να πω σε σχέση με τα όσα είπε η Κομισιόν τα Ήταν ε, γνωστός ο ρόλος της Συγκναλίνα για τη Λιθουανία. Η ίδια η Κομισιόν πριν από δύο χρόνια ή τρία έκανε μια αλλαγή του νόμου ούτως ώστε τα χρήματα για τον παροπλισμό να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την ε, δημιουργία εναλλακτικών πηγών ενέργειας στις χώρες αυτές. Δόθηκε αυτό το δικαίωμα και χρησιμοποιήθηκαν έτσι αυτά τα κονδύλια. Το ερώτημα μας που εγείρεται είναι γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια από τα διευθυντικά ταμεία, γιατί αυτά ενδείκνυνται για κάτι τέτοιο. Και ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση στο γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά για τον ε, παροπλισμό. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια από τα τα ταμεία, αλλά τα χρήματα αυτά για τον παροπλισμό πήγαν εκεί. Γιατί. Και τώρα εσείς κύριε Μαρινέσκου μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτή τη συζήτηση. Ουδέμια απάντηση στο ερώτημα της κυρίας ε, Γκρέσλε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει εν συντομία να απαντήσει. Πολύ σύντομα. Δεν αλλάξαμε τίποτα. Ήδη προβλεπόταν αυτό στις ε, συνθήκες ε, προσχώρησης. Τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και για τον παροπλισμό και για την μέτρα μειώσεως των αποτελεσμάτων του παροπλισμού. Ε, ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρινέσκου έχει το λόγο τώρα. Με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα κονδύλια των διαρθρωτικών ταμείων για αυτό το σκοπό. Γιατί Θέλει να απαντήσει ξανά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εκτός μικροφώνου. Η νομική βάση ήταν η αρχική βάση και τα χρήματα των εθνικών ταμείων χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον για συγκρίσιμα μέτρα όπως μέτρα για την αποδοτική χρήση της ε, ενέργειας. Ευχαριστώ. Το ελεκτικό συνέδριο έχει κάτι να προσθέσει. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε εκ νέου το λόγο. Το ερώτημα της ερητή μου κυρία Γκέστρα είναι πολύ δικαιολογημένο. Εξέτασε τον ευτικό συνέδριο την κατάσταση και συνεπέρανε ότι δυστυχώς οι, οι συνθήκες για την ένταξη ήταν πολύ γενικόλογες. Θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ποικιλοτρόπω. Και από τη στιγμή που δημιουργείται το πρόβλημα παροπλισμού ενό πυρηνικού αντιδραστήρια και κλεισίματό του, ε, διαθέτει ένα ευρύτατο, μεγαλύ, πολύ μεγάλο ποσό και προτιμάς να το χρησιμοποιήσει αυτό το ποσό για συγκεκριμένα μέτρα. Ε, ασφάλεια ενέργειας, ε, μέτρα μείωσης των συνεπειών κυρίως αν θες να τα χρησιμοποιήσει σαν ειδικό ταμείο, από ειδικό ταμείο αντί διαθετικά ταμεία. Το εξετάσαμε διεξοδικότατα. Δεν ήταν ξεκάθαρο από τη συνθήκη. Οπότε έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν λέει ότι έγιναν τα αιτήματα των χωρών και δαπανήθηκαν τα χρήματα. Αυτό εννοούσαμε. Η διαχείριση ανετέθηκε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανεκοδόμηση και Ανάπτυξη. Είπε η Τράπεζα: Υπάρχει το αίτημα, θα έρθει η έγκριση γιατί υπάρχουν οι πόροι. Και ποτέ η Τράπεζα δεν είχε το καθήκον να θέσει τον τελικό, να υλοποιήσει τον τελικό στόχο, τον αφοπλισμό. Απλώ ήλεγχε αν τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όσο προβλέπετο. Γι' αυτό ζήτησα και το λόγο. Εμείς συστήσαμε ως ελεκτικό συνέδριο ότι από τούδε και στο εξή τα μέτρα μειώσεως τα χρήματα παροπλισμού δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς μειώσεως των συνεπειών. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν άλλοι πόροι όπως τα διαθωτικά ταμεία. Και αν θα είναι διαθέσιμοι πόροι, αυτό εξαρτάται από τις χώρες αποδέκτες που θα τα χρησιμοποιήσουν και προβλέπεται στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο το πολιτέ, ότι αυτά τα διαθωτικά χρήματα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον κατά 20% για εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότητα της ενέργειας και αυτό θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στα μέτρα μείωση των συνεπειών. Επαναλαμβάνω εκ νέου ότι με τα χαράς να λάβουμε την απάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να τη δεχτούμε μάλλον ότι στο μέλλον τα χρήματα τα οποία θα προτείνετε εσείς στο νέο δημοσιονομικό πλαίσιο θα χρησιμοποιηθούν μόνο για παροπλισμό και όχι για μέτρα μειώσεως των συνεπειών πλέον. Αυτή είναι θετικότατη συνέπεια για το μέλλον, όχι για το παρελθόν, αλλά για το μέλλον. Και όσον αφορά και τη μελέτη του συγκητού σα και όσον αφορά και την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Υπάρχει κάποιος που θέλει να πει την τελευταία λέξη πριν δώσω το λόγο στον εισηγητή ο κύριος Μπαλσίτη, μετά ο κύριος Κάλφιν και μετά θα πρέπει να κλείσουμε γιατί δεν μα μένει κι άλλος χρόνος. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε και πάλι το λόγο. Η συνάδελφός μου, η κυρία Γκρέσλε, πραγματικά έθεσε ένα δικαιολογημένο και καλό ερώτημα. Γιατί δεν μπόρεσαν να αξιοποιηθούν τα κονδύλια από τα διορθωτικά ταμεία για αυτό το σκοπό. Οι πυρηνικοί σταθμοί υπήρχαν τότε σε τρεις χώρες μέλη που ε, σύμφωνα με μια πολιτική απόφαση έπρεπε να κλείσουν. Και για τις 25 χώρες μέλη τότε το 2004 ε, τα... έγινε η διανομή των κονδυλίων βάσει ενός συστήματος για την εκπαίδευση, για τη γεωργία ή για άλλους ε, τομείς ούτως ώστε να μπορούν να βοηθηθούν τα νεότερα μέλη. Και εάν ε, όντως θα μπορούσαν να εξαπηθούν τα διορθωτικά κονδύλια για το κλείσιμο των εργοστασίων, δεν θα έμεναν καθόλου πόροι για τους υπόλοιπους τομείς και αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αυτός ήταν ο λόγος που υπήρξε το τέταρτο πρωτόκολλο στις ε, συνθήκε ε, προσχώρησης και δεν το διαψεύδει η Επιτροπή, υπήρξαν ορισμένε υποχρώσεις Και ε, θα ήθελα να επαναλάβω και πάλι ότι πραγματικά εκτιμώ τη μεγάλη συμβουλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να βρούμε μία λύση η οποία να ικανοποιεί και τα τρία θεσμικά όργανα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπαλτσίτη. Πήρα uh, το λόγο στο τέλος της συζήτησης γιατί ήταν κάτι με το οποίο διαφωνώ τουλάχιστον από αυτά που μας είπε το Ελεκτικό Συνέδριο. Νομίζω ότι δεν είναι στη δικαιοδοσία του Ελεκτικού Συνεδρίου να εξετάζει, να κρίνει πολιτικές αποφάσεις. Επί μακρόν μπορώ να επιχειρηματολογήσω για την ανάγκη ύπαρξης μέτρων μειώσεως των συνεπειών και νομίζω αυτά τα επιχειρήματα εξετάστηκαν όταν υπεγράφησαν οι συνθήκες προσχώρησης. Και εκπλήσω με τα μάλα που ακούω τώρα ότι το ελεκτικό συνέδριο αφισβητεί τις συνθήκες προσχώρησης που είναι, είναι τμήμα τη βασική νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω το ελεκτικό συνέδριο θα πρέπει να μα ενημερώσει κατά πόσο η χρήση των χρημάτων ταιριάζει με τη νομική βάση. Και αυτό θα ανέμενα από το ελεκτικό συνέδριο. Διαφορετικά, το να γίνονται πολιτικέ δηλώσει από πλευρά του και να ξανανοίγει εκ νέου η συζήτηση, νομίζω ότι δημιουργεί προβλήματα. Έχω προβλήματα. Πράγματι, μπορούμε να συζητήσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο κατά πόσο θα πρέπει να αλλάξει η χρήση των χρημάτων στο μέλλον. Διότι όταν μιλάμε για παροπλισμό, θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι ακολουθούμε επίση και τι τεχνολογικέ επιταγέ, Αλλά αυτή είναι απόφαση που με ληφθεί εδώ. Και εγώ είμαι έτοιμο να συμμετάσχω στη συζήτηση. Σα ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά έχουμε μόνο πέντε λεπτά και πρέπει να διακόψουμε στη συνέχεια και θα πρέπει να ακούσουμε και τον εισηγητή. Αλλά μπορεί να αποφασίσει να αφήσει αυτά τα πέντε λεπτά για συζήτηση. Τι λέτε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Αφήστε την κυρία Γκλέσλε, σας παρακαλώ για ένα λεπτό. 30 δευτερόλεπτα, δεν χρειάζομαι ένα λεπτό. Ε, είναι μέλημα του ελεγκτικού συνεδρίου και πάντοτε μείναμε σε αυτό να εξετάσει το ζήτημα της αποτελεσματικότητας. Και αν τα κονδύλια του παροπλισμού χρησιμοποιήθηκαν για ένα άλλο σκοπό, θεωρώ ότι δεν είναι εντάξει Γι' αυτό ε, υποστηρίζω το, την, την παρατήρηση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Κρέσλε. Το ελεγκτικό συνέδριο θα μιλήσει για 30 δευτερόλεπτα ένα λεπτό. Ε, θα είμαι πολύ σύντομος. Καταρχήν θα ήθελα να στήσω να διαβάσετε την έκθεσή μας. Ποτέ δεν είπαμε ότι τα χρήματα δαπανήθηκαν με ένα μη σωστό τρόπο. Τα χρήματα δαπανήθηκαν σύμφωνα με τη συνθήκη προσχώρησης και το ερώτημα της ε, μελλοντικής ε, χρήσης των κονδυλίων ε, τίθεται εξή. Εάν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια κονδύλια για τον παραπλησμό μελλοντικά, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον παραπλησμό. Παρακαλώ διαβάστε την έκθεση. Και η οι μελλοντικές δαπάνες για το μετριασμό των επιπτώσεων θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από άλλες πηγές. Ποτέ δεν πάραμε τέτοιου είδου πολιτικές αποφάσεις προσπαθήσαμε να σας παράσουμε κάποιες αποδείξεις ώστε να μπορείτε εσείς να λάβετε τις δικές σας αποφάσεις επί τη βάση αυτών των αποδεικτικών στοιχείων. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μαρινέσκου, θέλετε να κλείσετε. Χαίρομαι πάρα πολύ που ενδιαφέρονται τόσοι πολλοί συνάδελφοι για αυτή την έκθεση. Ήθελα να σας θυμίσω μόνο για τη Λιθουανία ότι ε, είχε μόνο 1,67 δις ε, Σλοβακία 330 εκατομμύρια, Βουλγαρία 867 εκατομμύρια. Πάρα πολλά λεφτά και θα συμφωνήσω με την κυρία Γκρέσλε ότι είναι πάρα πολλά τα λεφτά και δεν αποκομίσαμε κάτι αντίστοιχο. Δεν εκδόθηκαν όλες οι άδειες παροπλισμού Η πάυση λειτουργίας δεν είναι μια αναστρέψιμη όπως θα έπρεπε και αν κάποιος επαναλειτουργήσει τον πυρηνικό αντιδραστήρα, κανείς δεν ξέρει αν θα είναι ασφαλής, διότι έχουν ήδη ε, παροπλήσει κάποια παραρτήματα. Δεν ξέρουμε καν αν θα λειτουργούν ε, ε, όπως πρέπει οι αντιδραστήρε αν επαναλειτουργήσουν. Δύο-τρία σχόλια ακόμη. Ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μα είπε ότι μέσα στην πρόταση της Επιτροπής αναφέρεται ότι θα διακοπεί το 2020 η χρηματοδότηση. Εν μέρη αληθεύει αυτό. Εμέσως αναφέρεται αυτό, δεν είναι σαφές. Αναφέρεται ότι τα προγράμματα θα ολοκληρωθούν το 2017, 2018 και 20 αλλά δεν υπάρχει ε, σαφής ε, αναφορά ότι αυτά είναι τα τελευταία κονδύλια που θα εκταμιεύσει η Επιτροπή. Και κάτι άλλο, μέσα πάλι στην πρόταση της Επιτροπής, προβλέπεται μία ενδιάμεση αναθεώρηση κατά την οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την δυνατότητα να τροποποιήσει το συνολικό κονδύλι για την ευθύνη. Ο κύριος Μπαλσίτης μας είπε ότι θα έπρεπε να φέρει την ευθύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα διαφωνήσω μαζί του. Η ευθύνη βάσει των δημοσιονομικών κανονισμών βαρύνει σαφέστατα τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ως θεματοφύλακα της συνθήκης έχει ως μοναδική ευθυνή να συνδράμει τα κράτη-μέλη και τίποτα παραπάνω. Για τη συνθήκη τώρα, αυτό που είπατε, αληθεύει αυτό ότι έχουμε τον παροπλισμό από τη μία και τη μητυγγύησον, τη μείωση των συνεπειών από την άλλη. Όμως, το ποσοστό που χρησιμοποιείτε τώρα για τα μέτρα είναι υψηλότερο του ποσοστού που αντιστοιχεί στον παροπλισμό. Αυτό αναφέρεται και στην έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και γι' αυτό πρότειναν και προτείνω και εγώ μελλοντικά τα κονδύλια που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τον ε, παροπλισμό, ώστε να πληρείται η πρώτη απέτηση, ένα λεπτάκι, ασφαλής λειτουργία δηλαδή, ε, του πυρηνικού σταθμού. Για τους διαγωνισμούς, όπως το θέμα της κυρίας Γκρέσλε, Ακριβώς γι' αυτό προτείνω ο επιθεώρηση της χρήσης των κονδυλίων στο μέλλον βάσει των δημοσιονομικών κανονισμών και να κάνουμε και ένα παραλληλισμό ανάμεσα στο στη χρήση αυτών των κονδυλίων, τον έλεγχο μάλλον της χρήσης των κονδυλίων του παροπλισμού και τον έλεγχο της χρήσης των κονδυλίων μέσα στα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων. Θα διαπιστώσετε πόσο πελώριες είναι διαφορές ανάμεσα στους δύο ελέγχους. Σα ευχαριστούμε κύριε Μαρινέσκο, ευχαριστούμε την Επιτροπή για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ευχαριστώ και τα μέλη τη Επιτροπή που συμμετείχαν ενεργά στη συζήτηση. 3 Μαου μέχρι τι 12 το μεσημέρι οι τροπολογίε, άρα η ψηφοφορία θα γίνει στι 29 Μαου στην Επιτροπή και η Ολομέλεια μπορεί να εγκρίνει την έκθεση βάσει της ειδική έκθεσης του ελεγκτικού συνεδρίου και της ε, έκθεσης κοντών Ιούλιο. Θα περάσω στο επόμενο σημείο, δηλαδή την έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη, σημείο 7, συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Θα ακούσουμε τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως όλοι γνωρίζετε πολύ καλά, οι διαπραγματεύσεις για το νομοθετικό πακέτο της μελλοντικής πολιτικής συνοχής λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα. Πολλές από τις διατάξεις που θα ισχύσουν στον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία. Ζητώ συγγνώμη τα πήγανα και έξω από την αίθουσα διότι μιλάει ο κύριος Σταυρακάκη. Επαναλαμβάνω κύριε Πρόεδρε, πολλές από τις διατάξεις που θα ισχύσουν στον κανονισμό για την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία περιλαμβάνονται στις γενικές διατάξεις του κανονισμού. Σε αυτό το στάδιο των διαπραγματεύσεων έχω υποβάλει ορισμένε τροπολογίε, τι οποίε τι έχετε όλοι στο φάκελό σα, που σχετίζονται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία και αφορούν τα εξή. Οι τροπολογίε που έχουν προταθεί στο άρθρο 7 αφορούν δύο ξεχωριστά ζητήματα. Η πρώτη τροπολογία στοχεύει στο να παρέχεται στα κράτη-μέλη που συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα του στόχου τη Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία η δυνατότητα να αναθέτουν σε έναν και μόνο φορέα την έκδοση της γνώμης για θέματα ισότητας. Με αυτόν τον τρόπο θα πετύχουμε σημαντική απλοποίηση. Η δεύτερη τροπολογία προτείνεται προκειμένου να αποσαφανιστεί η διαδικασία για την τροποποίηση ενός προγράμματος συνεργασίας, καθώς η πρόταση της Επιτροπής δεν αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα. Προκειμένου να πλουστευτεί και να αυθυγραμμιστεί ο κανονισμός Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, με τον κανονισμό για τις κοινέ διατάξεις προτείνω μια τροπολογία στο άρθρο 20 η οποία ορίζει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να μπορούν να έχουν την ελεκτική αρχή εντός του ίδιου φορέα με τη διαχειριστική αρχή υπό την προϋπόθεση ότι οι δύο αυτές αρχές είναι λειτουργικά ανεξάρτητες. Αυτό είναι κάτι που προτείνεται για τα άλλα ταμεία αλλά δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία οι ελεκτικές αρχές μπορεί να μην έχουν τα απαραίτητα δικαιώματα για την εξαγωγή ελέγχου στα διάφορα κράτη-μέλη. Συνεπώς, η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει την ύπαρξη μιας ομάδας ελεκτών με αντιπροσώπους από όλα τα κράτη-μέλη. Οι τροπολογίες στο άρθρο 23 αποσαφηνίζουν ότι οι αντιπρόσωποι αυτοί θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και να διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και επαγγελματική δυνατότητα. Επιπλέον, η ελεκτική αρχή θα εξηγεί στη στρατηγική ελέγχου η, παραλαμβάνω ότι πλέον η ελεκτική αρχή θα εξηγεί στη στρατηγική ελέγχου της τα μέτρα που λαμβάνει για το σκοπό αυτό. Τέλος, η τροπολογία στο άρθρο 25 παρέχει τη δυνατότητα να γίνεται χρήση ενός ενιαίου λογαριασμού για όλες τις ταμιακές ροές σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας. Κάτι τέτοιο θα πλουστεύσει τη διαχείριση και θα προσφέρει διαφάνεια στην παρακολούθηση του έργου. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να κάνω μια αναφορά στις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον κανονισμό των κοινών διατάξεων και να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής μας στα ακόλουθα. Ο κανονισμός των κοινών διατάξεων θεσπίζει κανόνες για την εξέταση των επιδόσεων του 2017 και του 2019 προκειμένου να εκτιμηθεί η επίτευξη των ενδιάμεσων στόχων που περιλαμβάνουν τα προγράμματα δεν είναι εντελώ σαφέ με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη απέτηση στον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, δεδομένου ότι εμπλέκονται διάφοροι παράγοντε. Οι συμβάσει εταιρική σχέση που εισάγονται με τον κανονισμό των κοινών διατάξεων καθορίζουν τι ρυθμίσει για την εξασφάλιση τη ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων με του στόχου τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020. Ωστόσο, ο κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία δεν αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερότητες των συμβάσεων εταιρικής σχέσης που προκύπτουν από την διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και τρίτων χωρών που έχουν διαφορετικές δομές διακυβέρνησης. Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Κανονισμού των Κοινών Διατάξεων, συγκροτείται μια επιτροπή παρακολούθησης που θα παρακολουθεί την εφαρμογή του κάθε προγράμματος. Τέτοια επιτροπή παρακολούθησης πρέπει να συγκροτείται και για τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Ωστόσο, η πρόταση τη Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη τι ιδιαιτερότητε του εν λόγω στόχου, ιδίω όσον αφορά τα δικαιώματα ψήφου λόγω των διαφορετικών συστημάτων στα κράτη-μέλη και στι τρίτε χώρε. Σε αυτό το σημείο, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε με να ολοκληρώσω την παρέμβασή μου, αναμένοντα με ενδιαφέρον τα σχόλια των συναδέλφων. Σας ευχαριστούμε κύριε Σταυρακάκη. Προτού αρχίσει η συζήτηση θα ήθελα να ακούσω και τον εκπρόσωπο, ότι είναι εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν υπάρχει κάποιος, εκπροσωπείται για αυτό το θέμα η Επιτροπή, παρακαλώ. Ναι. Ταυτόχρονα μας απασχολεί αυτό το θέμα. Περιμένετε 10 λεπτά ένα τέταρτο θα έρθει αρμόδιος από τη Γενική Διεύθυνση και μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τις ερωτήσεις και να ακούσουμε τις απαντήσεις σε ένα τεταρτάκι. Ωραία. Ας γίνει λοιπόν η συζήτηση, αν υπάρχουν ερωτήσεις, ε, σχόλια για την έκθεση του κυρίου Σταυρακάκη. Παρακαλώ κυρία Γκρέσλε. Μπορώ να ρωτήσω πού βρίσκονται ε, προβλήματα ε, σε σχέση με την ε, Γενική Διεύθυνση όπου δεν το θεωρεί αναγκαίο να παρέμβει. Μα θα έρθει, θα έρθει ο, ο, αρμόδιος από τη Γενική Διεύθυνση σε 10 λεπτά. Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Θα μπορούσατε εσείς ενδεχομένως να τοποθετηθείτε για αυτά που μας είπε ο κύριος Σταυρακάκης, όχι. Θέλετε να το λόγο τώρα, όχι. Κύριος Σταυρακάκης τότε. Τι... Κύριε Πρόεδρε, τι άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, thank you. Uh, λοιπόν, ε, θα αναφέρω μόνο ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Πάλι 3 Μαΐου, πάλι 12 η ώρα. Νομοθετική πρόταση και άρα καταθέτουμε τροπολογίες για την νομοθετική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στις 29 Μαΐου του 2012 θα γίνει ψηφοφορία στην Επιτροπή Κοντ. Κλείνει το σημείο και... Περνάμε στην έκθεση του κυρίου Βόγκαν κοινέ διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία και κατάργηση του κανονισμού 1083 ε, του 2006. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να υπενθυμίσω πρώτα απ' όλα στους ε, συναδέλφους ότι είμαστε στο στάδιο της αρχικής ανταλλαγής ε, απόψεων ε, στις 23 Απριλίου στην Επιτροπή μας έγινε αυτή η πρώτη ανταλλαγή απόψεων και συζητήθηκε το έγγραφο εργασίας που μελετούσε τα, τους μελλοντικούς κανονισμούς από πλευράς βεβαίως Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών και η δική μας οπτική γωνία αντιλαμβάνεστε ότι διαφέρει από αυτή άλλων επιτροπών Πρόκειται για ε, γνωμοδότηση νομοθετικού περιεχομένου και άρα οι τροπολογίε που καταθέτουμε κατατίθενται αυτόματα ε, στι ε, προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίση νομοθετικού περιεχομένου. Υπάρχουν κάποια βασικά ζητήματα που, στα οποία εδράζουν οι τροπολογίε που θα παρουσιάσω σήμερα στου συναδέλφου. Ε, Πρωτού περάσουμε στις ε, τροπολογίες, ε, θα δουν οι συναδελφοί ότι έχω ένα μικρό επεξηγηματικό σημείο μας στην αρχή της γνωμοδότησης, όπου διευκρινίζω τα περί κοινών διατάξεων και δημοσιονομικού κανονισμού. Φυσικά είναι στοιχεία που γνωρίζουν οι συναδελφοί, όμως ήθελα μόνο να διευκρινίσω κάτι σε σχέση με την προσέγγιση μου. Δηλαδή, έχουμε κάποιες τροπολογίες για το κεντρικό, το βασικό τμήμα και κάποιες άλλες τροπολογίες που αναφέρονται στις κοινέ ε, διατάξεις Common Provisions. Δεκαπέντε είναι οι τροπολογίες ε, που έχω εισηγηθεί. Δεν θα τις ε, διατρέξω μία-μία μπορούν να το κάνουν μόνοι του οι συνάδελφοι. Μετά από κάθε τροπολογία πάντω. θα δείτε μια μικρή σύντομη αιτιολόγηση που ευελπιστώ να διευκρινίσει την τροπολογία προ όφελο των ε, συναδέλφων. Δεν θέλω λοιπόν να υψέλθω σε λεπτομέρειε για τι 15 τροπολογίες. Ε, θα σχολιάσω μόνο το, τα επιμέρου κεφάλαια και πιστεύω ότι όλα είναι σημαντικά για την Επιτροπή μα. Υπάρχει το ένα που εξετάζει το θέμα της διαπίστευση ε, Επίσης βλέπουμε τα που που προσφέρουν τα κράτη-μέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκαθάριση και ε, λογαριασμών, ε, ερμηνεία των ε, κοινών διατάξεων, αναβολές, αναστολές, δημοσιονομικές διορθώσεις. Όλα αυτά τα επιμέρους σημεία είναι ιδιαίτερη σημασία για την Επιτροπή μας αλλά και για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τους ίδιους τους μελλοντικού κανονισμούς και για τα κράτη-μέλη που είναι οι δικαιούχοι και θα είναι οι δικαιούχοι μελλοντικά των ε, διαρθρωτικών ε, ταμείων. Στο τέλος έχουμε την τροπολογία 15 η οποία αναφέρεται στις πράξεις ε, κατεξουσιοδότηση. Αντί να πολλαπλασιάζονται οι τροπολογίες που όμως έχουν κοινό αντικείμενο, η ομάδα μου ε, συντηρητική αποφάσισε να ακολουθήσουν αυτήν την άγουσα σε μία τροπολογία να συνδυάζουν ε, με όλα τα θέματα που σχετίζονται με τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση. Αυτή είναι η τροπολογία 15. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο για την έκθεσή του διότι έχουν ήδη εκπονήσει έκθεση για τους μελλοντικούς ε, κανονισμούς για τα ευρωπαϊκά ταμεία. Ευχαριστώ τους συναντέλους που με βοήθησαν με τροπολογίες και σχόλια να συντάξω την έκθεσή μου. Ευχαριστώ και την ε, Γραμματεία για την ε, υποστήριξή της και τέλος... Να πω ότι περιμένω με ανυπομονησία τα σχόλια των συναδέλφων και τις τροπολογίες που έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν μέχρι τις 3 Μαΐου. Σας ευχαριστούμε κύριε Βόγκαν. Δυστυχώς αρμόδιος είναι ο ίδιος ε, άνθρωπος από την ε, αρμόδια Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ε, ήταν αρμόδιος και για την προηγούμενη έκθεση. Κατέφθασε από ό,τι βλέπω. Θέλετε να σχολιάσετε εντάχει εσείς κύριε Φάζακα από πλευρά του ελεγκτικού συνεδρίου για το θέμα 6 μέχρι να έρθει ο κύριος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλετε να πείτε κάτι εφόσον έχετε συντάξει και εσείς έκθεση. Δεν έχουμε άλλα σχόλια για το θέμα. Δεν είμαι και εισηγητής για το θέμα. Δεν έχω λεπτομέρειες. Είμαστε ικανοποιημένοι. Thank you. Και το εγκρίνουμε με τα χαράς. Thank Σας ευχαριστώ. Σχόλια από πλευρά συναδέλφων η κυρία Γκρέσλε. Ναι, πραγματικά θα το εκτιμούσα εάν μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση παρουσία τη αρμόδια Γενική Διεύθυνση. Θα ήθελα να παρακαλέσω όλου του συναδέλφου συζητητέ να συμπεριλάβουν ένα σημείο. Το Συμβούλιο προσπαθεί ούτε ώστε στο θέμα ε, για το πώς ε, γίνονται τα, λαμβάνονται τα στατιστικά δείγματα για τη διαπίστωση των σφαλμάτων ε, τα αστικά αυτά δείγματα δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τέτοιο δείγμα το οποίο είναι τυχαίο και βασίζεται σε κινδύνους. Ε, και αν δούμε, για παράδειγμα, στα γεωργικά ταμεία, ότι στο ένα δείγμα τελικά τα αποτελέσματα είναι χειρότερα από τη βάση της άλλης ε, δειγματοληψίας. Δηλαδή, άρα η ανάλυση των κινδύνων δεν είναι ε, αξιόπιστη. Ε, θα πρέπει κάτι να γίνει γιατί αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τελικά να μην μπορούμε να εγγυηθούμε μια αντιπροσωπευτικότητα βάσει του ποσοστού σφαλμάτων. Το Συμβούλιο ε, θέλει να υποβάλει τόσο στατιστικές όσο και μη στατιστικές μεθόδους. Δηλαδή, για παράδειγμα, να προσπαθήσει και αυτό θα μπορούσε να έχει ένα αποτέλεσμα να προσπαθήσει κανείς να υποβάλει σε έλεγχο μόνο ένα συγκεκριμένο τμήμα του προγράμματος. Κάτι το οποίο επίσης κατά την άποψή μου δεν είναι αξιόπιστο και δεν είναι αντιπροσωπευτικό όσον αφορά τα σφάλματα. Ε, γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν να παρακλέψω στους συναδέλφους να συμφωνήσουν το μη στατιστικό να διαγραφεί να υπάρχει δηλαδή μία δειγματοληψία με την ε, δυνατότητα να γίνονται οι αναλύσεις αυτές και να υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται μη στατιστικές ε, αναλύσεις. Ε, χρειαζόμαστε αυτό το ποσοστό σφαλμάτων, ούτε ώστε να υπάρξει κάποια πειθαρχία όσον αφορά την εφαρμογή. Δεν είναι δυνατόν να το ακυρώσουμε αυτό τελείως. Χρειαζόμαστε το περιθώριο των σφαλμάτων, του ποστό των σφαλμάτων. Uh, Ελπίζουμε. Θέλουμε τις παρατηρήσεις σας και τα σχόλιά σας. Κύριε Βόν, θέλετε να σχολιάσετε σύντομα, επειδή δεν βλέπω άλλο συνάδελφο να πάρει το λόγο και να κλείσουμε το, τη συζήτηση. Πολύ σύντομα, διότι νομίζω ότι αναφέρθηκε μόνο ένα στοιχείο, ότι η ίδια η έκθεση και οι τροπολογίες αναφέρονται στην προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο και αυτό ακολουθεί την προσέγγιση. Κρίμα που δεν είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκφράσει άποψη από αυτού. Μπορούμε να υποβάλουμε σχετικέ τροπολογίε. Ο υποφαινόμενο ή η κυρία Γκρέσλε, αν αισθανθούν ότι πρέπει να ενισχύσουμε, να προσαρμόσουμε συγκεκριμένο σημείο, να το κάνουμε μέσω τροπολογία. Uh, Ευχαριστώ. Δεν ζητάει άλλο το λόγο. Οπότε ανακοινώσω απλώ ότι η προθεσμία για τι τροπολογίε είναι η 3η Μαΐου, 3 Μαΐου, 12 το μεσημέρι. ψηφοφορία στην Επιτροπή θα λάβει χώρα στι 29 Μαΐου. Και εδώ ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο τη ημερήσια διάταξη. Επόμενο σημείο, το 5. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Τάμιο και αναστολή του 1081 του 2006, ε, πάυσης ισχύω αυτού, Κάταλη και ο συγγετής, ο κ. Γκάιερ, μήπως μπορεί να κάνει μια παρουσίαση εκ μέρου του. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα το ζήσετε αυτό πολύ συχνά σήμερα και αύριο. Δηλαδή να αναλάβω διάφορους ρόλους, διάφορες ιδιότητες. Ε, δεν τυχαίνει μόνο σε σένα, Ίγκε. Αυτό συμβαίνει όταν υπάρχουν μεγάλες αντιπροσωπείες που είναι πολύ απασχολισμένες. Η Καταλίνα αυτή τη στιγμή ακριβώς βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες και με παρακάλεσε να, να παρουσιάσω εκ μέρους της αυτή τη σύντομη γνωμοδότηση, το σχέδιο γνωμοδότησης. Όλοι κάπως ε, νομίζω υποφέρουμε όταν προσπαθούμε να ασχοληθούμε με τις διάφορες γνωμοδοτήσεις σε σχέση με τα διορθωτικά ταμεία γιατί ε, τελικά υπάρχουν παράλληλε διαβουλεύσει σε αυτή την Επιτροπή, στην Επιτροπή Προπολογισμού, στι διάφορε άλλε επιτροπέ, στην Επιτροπή Απασχόληση, στην Επιτροπή Περιφερειών κλπ. Ε, ή ταυτόχρονα γίνονται ε, διαβουλεύσεις για το γενικό κανονισμό και για τους ειδικούς κανονισμούς και δεν έχει ολοκληρωθεί ο δημοσιονομικός ε, κανονισμός, δεν έχουμε ε, κανένα δημοσιονομικό πλαίσιο, τελικά δεν έχει ολοκληρωθεί, γιατί θα πρέπει να γίνει αυτό στο τέλος. Άρα λοιπόν η γνωμοδότηση αυτή του Ιβαν τελικά πάσχει από αυτό το πρόβλημα ότι γίνονται αυτές οι διαδικασίες εκ παραλίλου, όλες οι βλέψεις εκ παραλίλου. Και έτσι λοιπόν χωλαίνει αυτό το σχέδιο διαγνωμοδότησης για το λόγο ότι ε, βρίσκονται εν εξελίξει διαβουλεύσεις και ο κανονισμός για τον προπολογισμό δεν έχει ολοκληρωθεί και επίσης δεν έχουμε και το γενικότερο πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι ε, συγητής ε, δεν μπορεί κάποιες επιφυλάξεις ε, όσον αφορά την υποβολή δικών του τροπολογιών σε ένα μεταγενέστερο χρονικό σημείο. και υποβάλλει κάποιες προτάσεις αυτές που δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να σας τις παρουσιάσω λεπτομεριακά. Thank Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ευτυχώς έχουμε τώρα εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να σχολιάσει την γνωμοδότηση. Ο κύριος Νόλεν Σένς της Γενικής Διεύθυνσης της Υπεύθυνης Απασχόληση ε, θα πάρετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο που παρουσίασε τη γνωμοδότηση. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για την πολύ περιεκτική σύντομη έκθεση για τον κανονισμό το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Όπως είπε και ο Σγκάερ, αληθεύει ότι κάποια θέματα δεν πρέπει να ειδωθούν απομονωμένα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Η πρώτη τροπολογία είναι μία που θα πρέπει να εξεταστεί σίγουρα εν ώψη και των άλλων προτινόμενων κανονισμών πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και άλλα σημεία είναι πολύ εύκολα, βοηθούν πολύ γιατί διευκρινίζουν το κείμενο. Το κάνουν καθαρό σαν κρίσταλο το τι μπορούμε να κάνουμε. Όπως η τροπολογία 3 η οποία ακολουθεί σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν άλλες όμως όπου θα πρέπει να εξεταστούν για να δούμε κατά πόσο συμβάλλουν στην απλούστευση του κειμένου ή όχι. Εμείς θέλουμε απλούστευση. Και στο συγκεκριμένο παράδειγμα για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θέλει ο εισηγητής να ετοιμάσει και κάποιες αλλαγές και με τα χαρά να έρθουμε σε επαφή με τον κύριο εισηγητή για να το κάνουμε αυτό. διμερός να συζητήσουμε το κείμενο. Αυτά και ευχαριστώ πολύ για το σχέδιο της γνωμοδοτήσεως. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος που θέλει να σχολιάσει τα όσα μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν δεν έχετε σχόλιο, κύριε Γκάιρ, θέλετε να πείτε κάποια πράγματα στο τέλος. Όχι. Οπότε τελειώσαμε αυτό το σημείο. Μισό λεπτό, κύριε Σταυρακάκη. Ο κύριος, κύριε Βον, είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εσά εξαρτάται να αποφασίσετε. Θέλετε να τους δώσουμε το λόγο. Ο οι συγητές αποφασίζουν. Okay, why not? Uh, <laughs> but first, uh, uh, I close item 5. Τελειώσαμε το σημείο 5. Προθεσμία υποβολή τροπολογιών της Μαΐου, ψηφοφορία στην Επιτροπή 29 Μαΐου. Οπότε ξαναπάμε στο σημείο 5. Κυρία Πρόεδρε, ο σκιώδης συγγετής μας κατέφτασε. Είναι η μέρα καθυστερήσεων. Ίσως θα μπορούσα να δώσω το λόγο για να αναφέρει κάποια σημεία προς συζήτηση. Αν υπάρχει χρόνο. Για ποιο σημείο ο συγητής, ρωτάει ο Πρόεδρος. Για ποιο σημείο. Έχουμε λοιπόν, δίνουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια σύντομη παρέμβαση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λυπούμε που δεν ήμουν εδώ όταν ξεκίνησε η συζήτηση του σημείου. Ήμουν σε άλλη συνεδρίαση. Μου είπαν ότι, ότι άλλαξε το σημείο συζητήσεως του θέματός μου. Τόσο αφορά το ETC, το θέμα είναι σχετικά με τα προτινόμενα ο συσχετισμό μεταξύ του κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και των διατάξεων για τις κοινέ διατάξεις σε σχέση με κάποια τα ζητήματα. Κάποια σημεία ήδη καλύφθηκαν όσον αφορά το Ταμείο Ευρωπαϊκή Στατική Συνεργασία, όσον αφορά τον κανονισμό με τι κοινέ διατάξει. Και τι προσπαθήσαμε να κάνουμε στον αφορά τον κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Λευκή Συνεργασία, να εισαγάγουμε συγκεκριμένες ρήτρε όταν αυτό ήταν αναγκαίο για να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες αλλά να μην επαναλάβουμε αν δεν χρειάζεται αυτά που αναφέρονται ήδη στις κοινέ διατάξεις και στον σχετικό κανονισμό όπως το άρθρο 116 που αφορά τις τροπολογίες 1, 5 και 6 πιο συγκεκριμένα. σχετίζεται και με τη διαδικασία για τα προγράμματα και τις τροπολογίες και το θέμα του διαχειριστικού φορέα και του ελεκτικού φορέα που θα έπρεπε να ανήκουν στο ίδιο πλαίσιο. Δεν το θεωρούμε ανάγκη αυτό να αναφέρεται γιατί καλύπτεται. Μετά, η τροπολογία που αφορά το άρθρο 25.1 είναι κάτι που δεν χρειάζεται. Προστίθεται στη διάταξη περιπληρώμων σε ενιαίο λογαριασμό, όπου υπάρχει και μια φράση που αναφέρεται σε έσοδα και έξοδα, που ίσως δημιουργεί σύγχυση. Και οι σχετικές διατάξεις ήδη βρίσκονται στον κανονισμό με τις κοινέ διατάξεις. Ευχαριστώ κύριε Σταυρακάκη, θέλετε να πείτε κάτι, όχι. Οπότε τελειώνουμε με αυτό το σημείο. Και πάμε στο σημείο 6 τώρα, όπου δεν ακούσαμε τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να δώσω το λόγο καταρχάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξανά ευχαριστώ, Πρόεδρε, για τη δυνατότητα που μου δίνετε να αναφέρω σε αυτό το θέμα. Στι περισσότερες περιπτώσεις, όσον αφορά τις προτάσεις κειμένου, βλέπουμε ότι ακολουθούν παρόμοια κατεύθυνση αυτή που θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν υπάρχουν ουσιαστικά προβλήματα να αναφερθώ στα μόνα σημεία που θεωρούμε ότι δημιουργείται πρόβλημα. Πρώτα απ' όλα στην τροπολογία 5 υπάρχει πρόταση επανεισαγωγή τη εγκρίσεω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Στρατηγική Ελέγχου. Προτείνεται στην τροπολογίε αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το σκέφτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το συμπερίλαβε στι δικέ προτάσει. Είναι κάτι το οποίο το εφαρμόζουμε στην ε, παρούσα πραγματική περίοδο και συνδέουμε την εξέταση του τι θα κάνουμε με τη διαδικασία πιστοποίησης με τη διαδικασία ελέγχου. Τι είδαμε, ότι δεν ήταν αποτελεσματικό από πλευρά κόστο να έχουμε συστηματική εξέταση εκ των προτέρων κάθε στρατηγική ελέγχου. Αυτό καλύπτεται επαρκώ από τι διατάξει που έχουμε στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα τι οποίε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει διαδικασία ελέγχου όταν το επιθυμεί. Άρα είναι θέμα ισορροπία. Να εξισορροπήσουμε τη διοικητική παρέμβαση με το κέρδο που επιτυχαίνουμε. Αναλύσαμε αυτά που έγιναν για την περίοδο 2013 και είδαμε ότι δεν υπήρχε καλή ισορροπία όσον αφορά προσπάθειες που κατέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το επιτυγχανόμενο κέρδος. Τροπολογία 7. προτείνεται συγκεκριμένη απέτηση για τι συμπεριλαμβάνεται σε αιτήσια έκθεση δραστηριοτήτων. Έχουμε επιφύλαξη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την αναφορά τη συγκεκριμένη σε κανονισμό του Συμβουλίου και του ε, Κοινοβουλίου το περιεχόμενο τη ετήσια εκθέσεω δραστηριοτήτων που αποτελεί εσωτερικό έγγραφο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Γενικού Διευθυντού. Και ουσιαστικά θα είναι κρίσιμο στοιχείο αυτό. Να αναφέρεται πώς δόθηκε ε, η έγκριση. Είναι σημαντικό, μεν, αλλά δεν νομίζουμε ότι πρέπει να αναφέρεται ρητά στον κανονισμό. Τροπολογία 15. Ρόλος του Ευρωπαϊκού Λεκτικού Συνεδρίου. Να εκφράζει την άποψή του στις κατεξουσιοδότηση πράξης. Επιφύλαξη. Δεν ξέρουμε κατά πόσο πρέπει να απαιτείται συστηματικά κάτι τέτοιο. Τελικό σχόλιο. Κάτι υπόθηκε όσον αφορά τη μη στατιστική δειγματοληψία. Είναι κάτι που προέκυψε από τη συζητή στο Συμβούλιο. Και αυτό σε σχέση με το άρθρο 116. Δημιούργησε δύο προβλήματα το 116. Το 116.1, εκεί πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι ελεγκτικέ αρχές θα πρέπει να καλύπτουν έλεγχο συστημάτων, του συστήματο και κάποιε επιχειρήσει. και θα πρέπει να ε, κρίνεται ποιο θα είναι το δέον δείγμα και αυτό θα κρίνεται κατά εξουσιοδότηση μέσω κατεξοδότηση πράξη. Έχει άλλη πρόταση στο Συμβούλιο τώρα από πλευρά Προεδρία. Η δειγματοληψία μπορεί να γίνει με στατιστική μέθοδο ή μη στατιστική μέθοδο. Και οι δύο μέθοδοι είναι ισότιμε. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέστησε σαφέστατο στι συζητήσει στο Συμβούλιο στι δύο συνεδριάσεις της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων ότι έχει πολύ μεγάλες επιφυλάξεις. Θεωρεί ότι δεν είναι δεδειγμένο αυτές οι δύο μέθοδοι δειγματοληψίε να είναι ισότιμε. Αυτό ίσω υπονομεύσει όλη την αρχή για ενίο έλεγχο αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει το μέσο να εναρμονίσει τον τρόπο δειγματοληψίας, ορισμού δειγματοληψίας, αυτό αμφισβητεί την αξιοπιστία από πλευρά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην γνωμοδότηση των εθνικών ελεκτικών αρχών και συνεπώ μπορεί αυτό να έχει σοβαρέ συνέπειε. Αυτή είναι η θέση στην οποία εμένει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού. Άρθρο 116, παράγραφος 5, που συνδέεται με αυτού. Υπάρχουν αλλαγές όσον αφορά τη διατύπωση της νομοδοτήσεως των ελεκτικών αρχών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε εκ νέου ανησυχίε επ' αυτού και αναφέρει ότι κατά την άποψή της και τα δύο ζητήματα συνδέονται άμεσα με τις συζητήσεις με θέματα άρθρο 56 του δημοσιονομικού κανονισμού και συνεπώς αυτά τα δύο σημεία θα έπρεπε να παραμείνουν στο περιθώριο και να περιμένουμε να δούμε τα τελικά αποτελέσματα των συζητήσεων όσον αφορά το άρθρο 56. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Μάρτιν. Και για τη συμβολή σα στι συζητήσει. Σκιώδη ηγητή του ΕΛΚ. Θέλει να πει κάτι. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε επειδή συνεργάστηκα με την ε, ε, Περιφερειακή Επιτροπή, με τον κύριο Βόγκενάου, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα. Καταρχήν, ε, συγγνώμη που καστέρισα λόγω συγκοινωνιακού προβλήματος, αλλά ευτυχώς μπόρεσα να φτάσω έγκαιρα. Ως ΕΛΚ συμφωνούμε απολύτως με, την, με τις τροπολογίες, καταρχήν τις γενικές ε, αρχές, το άρθρο 4 για τη δημοσιονομική διόρθωση που αφορά τα ελλείμματα επίσης στο σύστημα ελέγχου των χωρών μελών. Θα πρέπει να συμπεριληφθούν ε, και αυτά τα, αυτές οι ελλείψεις. Επίσης το άρθρο 5 που τονίζει τον ισχυρό ρόλο της Επιτροπής στους ελέγχους, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια, αν μια στρατηγική ελέγχου από την ίδια την Επιτροπή και βεβαίως αυτό μπορεί να συνεπάγεται ένα μεγάλο διοικητικό άχθος. Γι' αυτό ε, ίσως ε, κύριε το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να να συζητήσουμε κατά πόσο εδώ ε, δεν θα πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται κατόπιν ετήματος της Επιτροπής για να διενεργηθούν συνέχεια κάποια έλεγχοι. Και θα ήθελα να συζητήσω σχετικά με τον εισηγητή τώρα όσον αφορά την τροπολογία 15 για το άρθρο 137 που αφορά τα, τις δημοσιονομικές διορθώσεις που και κατά πάσα πρέπει να διατίθεται από εσά το ίδιο κεφάλαιο του προϋπολογισμού. Πράγματι θα πρέπει να συζητήσουμε κατά πόσο οι χώρες μέλη πράγματι στην περίπτωση αυτή ε, μπορούν να λάβουν χωρίς κυρός λίγο πολύ τα κονδύλια αυτά ή κατά πόσο τα διορθωμένα κονδύλια εμπέπτουν στη δίκηση της Επιτροπής και ε, προορίζονται σε ορισμένους τομείς διαρθωτικούς για παράδειγμα εκεί που υπάρχουν συγκεκριμένα καυτά προβλήματα και ε, στην περίπτωση αυτή να εκχωρείται μια ιδιαίτερη ευθύνη στην Επιτροπή. Επίσης το σημείο 4 που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, εν πάση περιπτώσει τα διορθωτικά ε, κονδύλια θα πρέπει να διανέμονται κάτω από μια κοινή, διοίκηση, κοινή διαχείριση. Ε, επίσης ε, το θέμα της ε, διαπίστευσης. Βεβαίω αυτό απαλλάσσει την Επιτροπή και μπορεί να εστιάσει τα κονδύλια σε ορισμένες χώρες που εμφανίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Αλλά θεωρούμε ότι είναι κάπως ανεπαρκώς διατυπωμένο, γιατί στην περίπτωση αυτή έχει το δικαίωμα παρέμβαση επιτροπής για αυτές τις χώρες μέλη, δηλαδή μπορεί να αναλάβει κάποια καθήκοντα ελέγχου. Και ίσως αυτό θα μπορούσε να διατυπωθεί πιο ξεκάθαρα στον κανονισμό. Και ένα τελευταίο σημείο, το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, όσον αφορά τις λεγόμενες δηλώσεις εξοπιστίας των χωρών μελών. Πιστεύω ότι εδώ χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια και η μεγάλη επιθυμία είναι οι χώρες μέλη να κοινοποιούν τα περιθώρια σφαλμάτων τους, να το κάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα και ε, να μπορούμε λοιπόν να το εξετάσουμε και εμεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι ίδιε οι χώρες λέει κουσίω να θέτουν στη διάθεσή μα τέτοια δεδομένα. Εγώ εκ μέρου του ΕΛΚ θα ήθελα να συζητήσω και πάλι το θέμα αυτό με τον εισηγητή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πίπερ. Θέλει η Επιτροπή να προσθέσει κάτι, δεν ξέρω, γιατί ε, και κάποια ερωτήματα. Εάν όχι, τότε το λόγο έχει ο κύριος Βον. Ευχαριστώ. Θα μπορώ να είμαι πάρα πολύ σύντομο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Σκιώδη Συγητή για τα σχόλιά του και την ευρύτατη υποστήριξή του. Έθεσε διάφορα ζητήματα που είναι λεπτομέρειε, αλλά δεν ξαφνιάζει κανέναν αυτό, διότι είναι τεχνικό το ζήτημα. Με τα χαράς λοιπόν να τα συζητήσουμε. Ε, όσο προχωρούμε στην εξέταση και λαμβάνουμε και τις τροπολογίες μέχρι τις 3 ε, ε, Μαΐου. Μπορώ να συζητήσω μαζί του και με άλλους συναδέλφους όλα αυτά τα ζητήματα. Σε σχέση με τα, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα τους ευχαριστούσε επίσης. Μπορούμε να δούμε τα δύο-τρία σημεία που έθιξαν Θυμάστε την τελευταία συζήτηση που κάναμε σε μια προηγούμενη συνεδρίαση επί του εγγράφου εργασίας. Ε, το θέμα είναι να διασφαλίσουμε ότι θα πλουστευτεί η διαδικασία για όλους, όχι μόνο για τα κράτη-μέλη ταυτόχρονα όμως. Η ευθύνη ευθύνη για, τη, όλα αυτά τα κονδύλια και για την εκτέλεση των προγραμμάτων, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ε, ε, ότι βαραίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουμε καταθέσει σχετικές τροπολογίες για την διαπίστευση. Ε, νομίζω ότι αν επιλέξουμε την ε, λύση των διαχειριστικών ε, αρχών είναι μεν ε, θετικό, αλλά η τελική ευθύνη πρέπει να βαραίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά τα πράγματα και θα τα ξανασυζητήσουμε και θα καταθέσουμε σχετικές τροπολογίες. Ε, Πρόεδρος, ο ελεγκτικός συνέδριο θέλει να κάνει ένα τελευταίο σύντομο σχόλιο. Ευχαριστώ. Ε, Ξανά το θέμα. Δεν ε, θέλησα πρόμισα όρο να παρέμβω για το ίδιο θέμα, διότι θα θυμάστε ότι πριν από δύο μήνες σας παρουσίασα την γνωμοδότηση του ε, συνεδρίου που καλωσόρισε ο εισηγητής σας, κύριος Βούν, και εφόσον δεν υπήρξαν σχόλια θεώρησα ότι δεν συνέτρεχε λόγος για να παρεύουμε. Τώρα όμως ακούσαμε και τον Σκιώδη Σιγητή, ακούσαμε και τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχω κάποια πράγματα να πω. Πρώτον, Εκτιμούμε ιδιαίτερως ε, την έκθεση του κυρίου Βον, κυρίως ως προς δύο σημεία της, ε, που αμφισβητεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τροπολογίες 7 και 15 συγκεκριμένα εκεί επαναλαμβάνει κάποια στοιχεία από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και χαίρομαι που απάντησε ορθά στι ερωτήσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, τι σημαίνει η τροπολογία 7, ότι η ε, ίστατη ευθύνη, η τελική ευθύνη βαραίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, ο ελεγκτικό ρόλο τη Επιτροπή στη διαδικασία διαπίστευση πρέπει οπωσδήποτε να ληφθεί υπόψη. Στη 15 υπάρχουν τουλάχιστον 7 παράγραφοι που έχουν ε, το ίδιο αντικείμενο, δεν χρειάζεται το να το σχολιάσω αυτό. Θα ευχαριστήσω μόνο τον εισηγητή για τις προτάσεις του και την Επιτροπή σας. Ε, ευελπιστώ ότι θα ε, ληφθούν υπόψη οι προτάσεις του ε, στον επόμενο κανονισμό. Σας ευχαριστούμε όλους για την υπομονή σας και τη συμμετοχή σας στην συνεδρία. Συνεχίζουμε αύριο στις 7. coordinators meeting is at